Θα ήθελα σήμερα να απευθύνω μια στοργική σκέψη στην ε, Νικόλ Φοντέν που μας άφησε πριν από λίγες μέρες μετά από μια, ένα μακρύ πολιτικό βίο αφιερωμένο στην υπηρεσία της κοινωνίας και στον αγώνα για τα ιδανικά της ανάμνηση γεμάτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη. Εξελέγει για πρώτη φορά το 1984. Ήταν εξέχον μέλος της ε, συνελευσής μας ε, για 23 χρόνια με μία μόνη διακοπή δύο ετών όπου διατέλεσε υπουργό στη Γαλλία. Όλα αυτά τα χρόνια απέκτησε μια βαθιά γνώση του Κοινοβουλίου και του πολιτικού και θεσμικού ε, περιβάλλοντος της Ένωσης και εργάστηκε ε, διαρκώς για την ανάπτυξη του θεσμού μας. Εργάστηκε με πάθος για την εδραίωση της διαδικασίας συναπόφασης και για την ε, αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Της χρωστάμε πάρα πολλά. Στις 20 Ιουλίου 1999 20 χρόνια μετά από την πρώτη γυναίκα της Σιμών Βέλη ε, ε, ορίστηκε πρόεδρος της συνέλευσής μας. Μια πραγματική ομόνια. Ε, ενωμένη στην διαφορά αυτό της το σύνθημα που μετετράπησε δικό μας σύνθημα ήταν αυτό που τη χαρακτήρισε. Αυτή η σελίδα της ιστορία μας ε, είναι πολύ σημαντική και αυτό το σύνθημα, αυτό το ρητό εκφράζει τη σκέψη και το νήμα της πολιτικής της δράσης. Βεβαίως είμαστε διαφορετικοί και οι διαφορές μας μας, μας εμπλουτίζουν. Αποτελούν ε, μια κοινή ευρωπαϊκή ε, κουλτούρα ε, τριών χιλιάδων ετών. Ναι, κάποιες φορές έχουμε διαφορετικά συμφέροντα, αλλά έχουμε τις ίδιες, μοιραζόμαστε τις ίδιες κοινέ θεμελιώδεις αρχές και μόνο ενωμένοι μπορούμε να τις πυροσπιστούμε και να τις προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιο ήταν το πνεύμα της όταν στο όνομα του Κοινοβουλίου υπέγραψε το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων πριν από 18 χρόνια. Ήταν πεπισμένη ότι η δική μας ε, κοινοβουλευτική συνέλευση θα πρέπει παντού στον κόσμο να διαδώσει τις αξίες αυτές, ειδικά στα μέρη όπου η δημοκρατία παραβιάζεται ή ε, δυσκολεύεται να επικρατήσει. Γι' αυτό και ε, είχε μια ιδιαίτερη ματιά για την Αφρική. Είμαστε σε ένα μέρος του κόσμου όπου η θανατική ποινή δεν ισχύει. Μόνο θα πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας όταν φυλακίζονται δημοσιογράφοι, όταν οι γυναίκες στερούνται την ελευθερία τους, υπόκεινται σε βία. Πρέπει να λειτουργήσουμε ως φάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή ήταν η βαθιά πεποίθηση της Νικόλ Φοντέν. Μόλις εξελέγει πρόεδρος ε, του Ευρωκοινοβουλίου το 1999, η Νικόλ Φοντέν επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη εγκύτητα με τους Ευρωπαίους πολίτες. Και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στο κατάπαυστο έργο της, το οποίο εκφράζεται μέσω του έργου της, αλλά και μέσω της τακτικής και εντατικής της παρουσίας επιτόπου, κοντά στους πολίτες. Στη διάρκεια της Προεδρίας της θα ε, επισκεφθεί ε, όλες τις χώρες για πάνω από 100 διασκέψεις και παρεμβάσεις. Αυτή η παρουσία, ε, το ότι ήταν κοντά στους πολίτες, συνοδευόταν από μια εξαιρετική ικανότητα συνομιλίας και ακοής ε, προς τους άλλους που ήταν καθοριστική τη στιγμή κυρίως της έγκρισης των νέων νομίσματος ενώ ε, αυτό είχε προκαλέσει πολλούς φόβους στους Ευρωπαίους. Να θυμίσω επίσης την έκθεση Φοντέν με την οποία αποφασίσαμε να χορηγήσουμε βοήθεια στις ε, αδελφοποιήσεις ανάμεσα σε δι... ευρωπαϊκούς δήμους μια μικρή χειρονομία που επέτρεψε την προσέγγιση και την αμοιβαία επαφή και γνωριμία ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτή η αρχή της εγκύτητας είναι, και της γειτονίας είναι ουσιαστική και σήμερα. Η Νικόλ Φοντέν ήταν μια διορατική και θεραλέα πρόεδρος, ενώ οι Ταλιμπάν ε, διέλυαν το Αφγανιστάν, εκείνη κάλεσε τον ε, τον ε, καπετάν Μασούντ στις Βρυξέλλες ε, παρά τις αντιδράσεις ε, καθώς και τον πρόεδρο της Παλαιστινικής Αρχής και της Κνέσεντ. Ήταν μια σπουδαία στιγμή για στο Κοινοβούλιο. Στη διάσκεψη κορυφή τη Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000 κατάφερε να πείσει τον Τόνι Μπλερ ότι ήταν ανάγκη να υπογραφεί ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανακτήρια ομιλία τη το 1999 έλεγε Σήμερα πρέπει επιγόντως να δώσουμε νόημα στην Ένωση. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από αυτή την άποψη. Τώρα είναι δική μας σειρά να συνεχίσουμε το έργο της ε, διακεκριμένης μας αυτής συναδέλφου που ήξερε να μιλά στον κόσμο. Πρέπει να ξυπνήσουμε τον ενθουσιασμό, να, να αναζωογονήσουμε αυτό το αίσθημα του ανήκειν σε αυτό το μεγάλο ε, όραμα. Στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Νικόλ, για αυτό που ήσασταν, για το πάθος, το θάρρος, που σηματοδότησαν την εργασία σας στην υπηρεσία των πολιτών, στη διάρκεια της ζωής σας και όπως τα λέγατε συχνά, για να ολοκληρωθεί αυτή η ένωση. Ε, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Βέμπερ για τέσσερα λεπτά, ώστε να μιλήσει για την Νικόλ Φοντένα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στα αγγλικά ο κύριος Βέμπερ, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε συντετριμένοι από την απώλεια της Νικόλ Φοντένα τα πιο ειλικρινή μα συλληπιτήρια θέλουμε πρώτα απ' όλα να στείλουμε στην οικογένειά τη και του φίλου τη. Η οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη του. Και ένα ειλικρινή φίλο, μια ειλικρινή φίλη που ήταν παραστάτη στο πλευρό μα περίπου 23 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, η Νικόλ Φοντέν ήταν πάρα πολύ ενεργή σε θέματα Πολιτική ε, εκπαίδευση και παιδεία. Ήξερε ότι οι κοινωνίε μας χρειάζονταν αξίες και επίσης γνώριζε ότι το κλειδί για να αποκτήσει κανείς αξίες είναι η παιδεία. Αυτό είναι για ένα φάρος της χριστιανοδημοκρατία. Η Νικόλ Φοντέν υπήρξε σπουδαία χριστιανοδημοκράτη. Και επίση ήταν και ακρεφνινό πεπισμένη Ευρωπαία. Ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα πόσο σπουδαία γυναίκα και πόσο δυνατή. Μόλις πρόσφατα η Νικόλ Φοντέν μας απέφθινε μια έκκληση για να ξαναλανσάρουμε την Ευρώπη. Μας είπε να ξανακάνουμε την Ευρώπη ένα εγχείρημα το οποίο θα ονειρεύονται και θα οραματίζονται οι πολίτες ας το υλοποιήσουμε αυτό στη μνήμη μιας μεγάλης σπουδαίας γυναίκας, μιας δυνατής, μιας χριστιανοδημοκράτης και μιας ε, πεπισμένης Ευρωπαίας. Σας ευχαριστώ. Προφανώς ο Πρόεδρος Βέμπερ υπενθύμασε εξ ονόματος όλων των πολιτικών ομάδων ε, την ε, φίγουρα της Νικόλ Φοντέν όπως έγινε και ε, για τη Σιμών Βέιλο και Φορφόρχα. Και τώρα στηρίσουμε ενός λεπτού σιγή τη μνήμη της. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Πέτερινγκ, ο οποίο θέλησε να παρευρεθεί σήμερα για να υπενθυμίσουμε την Νικόλ Φοντέν σε όλου. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, από την